από την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκουν και βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ και την κυρία Σβένσον, η οποία έλαβε μέρος στις εκλογές του Προέδρου και για όλες τις συζητήσεις που είχαμε μαζί. Για όλους τους συναδέλφους μας και ιδίως στον αναφερόμενο στον Μάριο Μάουρο και τον Γκράχαμ Βότσον, οι οποίοι ήταν προηγουμένως υποψήφοι και απεσύρθησαν για να διατηρήσουν την ενότητα του σώματος, Ξέρω πόσο σημαντικό ήταν αυτό, ιδίω για σένα Μάριο Μάουρο. Ξέρω πόσο σημαντικά ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα για σένα. Στη χώρα μου γεννήθηκε το κίνημα της και ένα μεγάλο κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό έγινε πραγματικότητα χάρη στις προσπάθειες και του ε, Ιωάννου Παύλου του Δεύτερου. Και Γκράμ, εσύ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να αλλάξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών μας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, γιατί οι πολίτες μας όλο και περισσότερο βρίσκονται σε μια κατάσταση αδιαφορία. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση πραγμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, κύριε υψηλέ εκπρόσωποι του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, <clears throat> σήμερα είναι 14η Ιουλίου, είναι η Εθνική Εορτή της Γαλλίας, είναι η επέτειος της Γαλλικής Επανάστασης συγχρόνως. Θέλω να ευχηθώ ε, ευτυχισμένη εθνική εορτή στους Γάλλους συναδέλφους μας και, και το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης βασιζόταν σε τρεις λέξεις. Ελευθερία, αδελφότητα και ισότητα. Σήμερα είναι μια συμβολική ημέρα. Ως εκπρόσωπος μιας χώρας της Κεντροανατολικής Ευρώπης θέλω να καταθέσω και προς όλους τους ευρωβουλευτές τη δική μου μαρτυρία για την ευθύνη που σημαίνει για μένα η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν νεότερο ήθελα να είμαι βουλευτή στην Πολωνική Βουλή τη στιγμή που η Πολωνία ξαναβρίσκεται τη δημοκρατία. Τώρα αναλαμβάνω το αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα άπιαστο όνειρο για μένα στο παρελθόν. Αυτό όμω δείχνει πόσο έχει αλλάξει η Ευρώπη μας. Νομίζω ότι η επιλογή του ατόμου μου ω πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι και ένα μήνυμα προ τι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Προ την Εστονία, τη Λιθουανία, τη Λετωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία και μια απότηση φόρου τιμή προ τα εκατομμύρια των πολιτών μα που δεν υποτάχθηκαν σε ένα <clears throat> εχθρικό ολοκληρωτικό σύστημα. Νιώθω ότι εκπροσωπώ το σύνολο των πολιτών από τις χώρες αυτές. Πριν από 20 χρόνια, το 1989, η Σολντανόσκ επέτυχε το στόχο της να υπάρχει μια ελεύθερη και δημοκρατική Πολωνία. Και αυτό ήταν η αρχή του τέλους για, την... για το σιδηρούν παραπέτασμα και για την καταπίεση των χωρών της Κεντροανατολικής Ευρώπης. Εμείς τότε βρισκόμασταν από την άλλη πλευρά του σιδηρούς του σιδηρού παραπετάσματος, αλλά μας βοηθήσατε κι εσείς με τις δικές σας προσπάθειες και με την υποστήριξή σας και καταφέραμε τελικά να επιτύχουμε το στόχο μας. Έτσι καταφέραμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Εδώ και πέντε χρόνια οικοδομούμε από κοινού μια κοινή Ευρώπη. Δεν είμαστε πια εμείς και εσείς, είμαστε όλοι εμείς. Είναι η δική μας Ευρώπη, η, Ευρώπη, η κοινή Ευρώπη που μας συνενώνει όλους. Αναφέρθηκα στο θέμα της ευθύνης μας. Όλοι μας έχουμε ένα τμήμα της εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η εξουσία είναι κυρίως η ευθύνη ενώπιον των πολιτών μας. Εγώ αισθάνομαι βαθιά αυτή την ευθύνη με την οποία μας έχουν επιφορτήσει οι πολίτες της Ευρώπης. Θα πρέπει να είμαστε θεματοφύλακες της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουν οι πολίτες της Ευρώπης από εμά να δείξουμε τον δρόμο εξόδου από την οικονομική κρίση. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, πρέπει να εργαστούμε, πρέπει να δώσουμε πρώτη έμφαση στην ανάκαμψη της απασχόλησης. Οι πολίτες μας θέλουν να έχουν τη βεβαιότητα ότι θα έχουν μια θέση εργασίας επίσης, ότι θα έχουν και την ενεργειακή ασφάλεια, θα μπορούν να έχουν φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Επίσης οι πολίτες μας θέλουν να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Ξέρουμε ότι πρέπει να αναχαιτήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα στο κλίμα του πλανήτη μας που έχουμε δει ήδη στην Αφρική, στην Ασία κτλ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση και την εταιρική σχέση με τις χώρες της Μεσογείου, τη νότια Όχθη Μεσογείου, την στρατηγική <clears throat> σχέση με τις χώρες της Λανική Αμερικής, με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τις άλλες διεθνεί δυνάμεις στο Διεθνέ τερέμα. Για να προχωρήσουμε λοιπόν είναι απαραίτητη για μας η συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα πρέπει να οργανωθούμε, να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από 30 χρόνια εξελέγει για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεσες και καθολικές εκλογές. Η πρόεδρος του ήταν τότε μία γυναίκα, μία Γαλλής, η Σιμών Βέη. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι και οι γυναίκες στην Ευρώπη θα πρέπει να ζουν σε συνθήκες ισότητες, να μπορούν και στο δημόσιο χώρο να δρούν σε ίσο επίπεδο με τους άνδρες και στον επαγγελματικό και στον πολιτικό χώρο, χωρίς να απαρνηθούν τη μητρότητα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, η πρόκληση της ελευθερίας, της ειρήνης και της ευμάρειας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με τρόπο αποτελεσματικό, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μονάχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι πια σε εθνικό επίπεδο μετά από 30 χρόνια. Αυτή είναι και η πρόκληση που αντιμετωπίζει το, Εθνικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί μου συνάδελφοι. Τα... Τις λεπτομέρειες του προγράμματός μου ως Προέδρου για τα επόμενα 2.5 χρόνια θα σας τα παρουσιάσω το Σεπτέμβριο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά τώρα θέλω να αναφερθώ στον προκάτοχό μου, τον Hans Gert Pöttering. Προσπαθώ να σε βρω, Hans Gert, ήταν μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή. Γνωριζόμαστε εδώ και δεκαετίες. Σήμερα μου έδωσε τη σκητάλη και μου παρέδωσε το υψηλότερο αξίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξ όλων των συναδέλφων μου θέλω να σε ευχαριστήσω. Νομίζω ότι κατάφερε να αποκομίσει τεράστια εκτίμηση όλων εξ του θεσμικού μα οργάνου. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την τεράστια πολιτική σου κουλτούρα και την τεράστια πολιτική σου ποιότητα ω Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Na pamiątkę, na pamiątkę. Ως ενθύμημα θα σου ένα αγαλματάκι της ε, Αγίας Βαρβάρας, της ε, προστάτηδος των ανθρακορίχων από τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, από τη Σιλεσία. Και σου εύχομαι και κάθε επιτυχία για το μέλλον και σε ευχαριστώ και πάλι εκ βάθους καρδίας. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Ιωσέφ Τόλ το λόγο. Président, ce n'était δεν προβλεπόταν κύριε Πρόεδρε, αλλά για μένα είναι μεγάλη χαρά και για ολόκληρο το Κοινοβούλιο, γιατί για πρώτη φορά στο Κοινοβουλίο δεν έχουμε Ευρώπη της Ανατολής ή της Δύσης, Δυτική ή Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε έναν Πρόεδρο ο οποίος εκπροσωπεί την ενότητα. Αυτή είναι η ενότητα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπες και πριν, φίλε Ζέρζι Μπούσεκ, αυτή είναι και η ευθύνη μας. Και αν μπορέσουμε στα επόμενα δυόμιση χρόνια της Προεδρίας σου να ξεχάσουμε την Ευρώπη, την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη και να μιλάμε για μια ενιαία Ευρώπη, αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Αυτό σου εύχομαι και τα επόμενα δυόμιση χρόνια της θητείας σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντόλ. Ο κύριος Σούλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θέλω να σε συγχαρώ εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδος για την εκλογή σου. Εμείς υποστηρίξαμε την εκλογή σου και θέλω να καταγραφεί ότι Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις ιστορικές στιγμές και τα ιστορικά γεγονότα, αλλά τολμώ να πω ότι η εκλογή σου στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μια ιστορική στιγμή. Γιατί βρισκόμαστε 20 χρόνια μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και πέντε χρόνια μετά από την προσχώρηση της δικής σου χώρας και πολλών άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά είναι μια διαδικασία που ήδη ξεκίνησε σαν πρωθυπουργό της χώρας σου με τις διαπραγματεύσεις ε, ένταξης της Πολωνίας. Αλλά βρισκόμαστε 20 χρόνια μετά από το ξεπέρασμα της ε, διέρεσης της Ευρώπης σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα 20 χρόνια μετά από το ξεπέρασμα της σταλινικής δικτατορίας που χρειάστηκε να ζήσετε 40 χρόνια περισσότερα από ό,τι έζησε τη δικτατορία το δυτικό τμήμα της Ευρώπης με τους φασίστες και τους ναζιστές. Με το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει παρουσία Πολωνών, Τσέχων, Ούγγρων Ευρωβουλευτών μαζί με τους ε, Γερμανούς, τους Αυστριακούς, τους Ιταλούς, τους Πορτογάλους κτλ. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι μαζί σε ένα κοινό κοινοβούλιο και σε μια ελεύθερη εκλογή μπορούμε να αναγορεύσουμε ένα εκπρόσωπο της Σολινταρνόσκ, έναν πρώην Πρωθυπουργό της Πολωνίας, στην κορυφή στο ύπατο αξίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό για μένα αποτελεί ένα πραγματικά ιστορικό γεγονότο και δείχνει ότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη ήπειρος η οποία περιλαμβάνει 27 κράτη και πράγματι αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται αυτό το όνειρο της Ευρώπης, το όνειρο της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Δεν είναι πλέον μονάχα ένα όνειρο, αλλά είναι μια ενεργή πραγματικότητα, κάτι που πετύχατε κι εσείς στη δική σας πολιτική ζωή και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι αξίες οι οποίες υπερνίκησαν τη δικτατορία σε όλη την Ευρώπη έχουν κερδίσει και αυτές είναι οι αξίες οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύουν και την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με όλα αυτά θέλω και πάλι να σας συγχαρώ εκ βάθους καρδίας. Γιάννη Σιμπούζεκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σούλτ, το λόγο έχει ο κύριος σας ε, συγχαίρω κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια από την ε, δική μου ομάδα, Φιλελευθέρων και Δημοκρατική, για την εκλογή σας και μπορώ να σας πω ότι έχετε την πλήρη υποστήριξη της ομάδας μας για τα επόμενα χρόνια της εργασίας σας. Της εργασίας σας που κατά τη γνώμη μου σημαίνει να δημιουργηθεί ε, μια πιο ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, θα είναι πολύ κοινοτική γιατί γινόσαστε πρόεδρο σε μια δύσκολη στιγμή. Πρέπει να επικυρωθεί η συνθήκη τη Λισαβόνα, να υπάρχει μια ενιαία στρατηγική κατά τη ε, οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Και αυτό το δύσκολο έργο έχετε να τον αντιμετωπίσετε με πλήρη υποστήριξη δική μα ομάδα και πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πίσω σα μια μεγάλη υπερευρωπαϊκή πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. το μόνο αίτημα που έχουμε είναι αυτή την πλειοψηφία που έχετε, που είναι υπέρ της Ευρώπης, να τη χρησιμοποιήσετε για να προχωρήσετε με την Ευρώπη και να πείτε ό,τι έχετε να πείτε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που γνωρίζετε τόσο καλά όπως το γνωρίζω και εγώ. Και ελπίζω εκεί να είσαστε η φωνή μας για να υπάρχει και εκεί περισσότερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Χάμς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα εξ νόμου τη ομάδα μα να συμφωνήσω με τα συγχαρητήρια των προληψάντων. Σημεριζόμαστε την χαρά για την στιγμή αυτή και θεωρώ ότι κάπω ε, ήσασταν περιοδικά τριοπαθή όταν είπατε ότι είναι μια τιμή να λάβετε αυτή, αυτό το αξίωμα σήμερα είναι μια ε, τιμή και για μας, ε, τουλάχιστον από πλευρά της δικής μας ομάδας, ε, ότι σας έχουμε ως πρόεδρο και πιστεύω ότι πραγματικά με όλη σας την πολιτική ζωή αξίζεται αυτό που αναλαμβάνετε σήμερα. Ε, που, ε, υποθέτουμε τις ελπίδες μας σε εσάς. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσον σε δυόμιση χρόνια θα είναι δυνατόν αυτό που χωρίζει ακόμα την, στην Ευρωπαϊκή Ένωση την Ανατολή από τη Δύση, αλλά ε, φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε εσείς επικεφαλής του σώματος να ενδυναμώσετε τις γέφυρες μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ε, θα ήθελα ιδίω οι συνάδελφοι από την Δυτική Ευρώπη να καταλάβουν καλύτερα ότι η Πολωνία βρίσκεται στο κέντρο της Επίρου μας ότι προέρχεστε από μια χώρα στο κέντρο της Επίρου και ότι η εργασία προς Ανατολάς θα πρέπει να είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι ήταν μέχρι στιγμής. Εσείς έχετε τις καλύτερες προϋποθέσεις γι' αυτό. Χάρηκα που είπατε ότι θα πρέπει να αναζητήσετε να είσαστε πλησίον του πολίτη. Αυτό είναι κάτι που εμείς ως πράσινοι θα το υποστηρίσουμε πάντα. Ένα είναι να ενδυναμώσουμε την Ευρώπη προς τα μέσα, το άλλο είναι να σκεφτούμε την Ευρώπη πιο μεγάλη και τώρα που σας γνώρισα πολύ καλά θα ήθελα να σας πω ότι όταν είχατε την πορτοκαλιά επανάσταση πήγα στους δρόμους του Κιέβου και σας γνώρισα σαν ένα τολμηρό πολιτικό. Και θα ήθελα να πω ότι ας μην ξεχάσουμε την Ουκρανία στον προσδορισμό μας προς Ανατολάς. Ελπίζουμε και εκεί να υπάρχουν καλύτεροι καιροί. Και αυτό που προσωπικά εγώ θα ήθελα θα ήταν εάν ε, ε, γίνουν, όταν γίνουν η ευρωπαϊκή το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που θα γίνει και στην Ουκραίνα, ας ε, πάμε μαζί να δούμε κάποια από τα παιχνίδια αυτά. Σας Ευχαριστούμε κάθε επιτυχία συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Καλώ τον κύριο που να πάρει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανάληψη της Προεδρίας και να καλωσορίσω το γεγονός ότι στα σχόλιά σας αναφερθήκατε στην ιστορία καθώς και άλλοι. Αλλά φαίνεται ότι είστε κάποιος ο οποίος αξιολογεί ιδιαίτερα τις ελευθερίες, την ε, ε, ελευθερία λόγου, αλλά και την αλλαγή και τη μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Και το σώμα αυτό πρέπει να αλλάξει και να δεχτεί τις μεταρρυθμίσεις της Ευρώπης. Εσείς έχετε μια ιστορία για την οποία είσαστε υπερήφανος μετά το 80 και τη Solidarnosc όταν εντάξατε και την Πολωνία στο ΝΑΤΟ και μετά αρχίσατε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε λοιπόν να προωθήσετε πολλών ειδών διαπραγματεύσεις και θα θέλαμε να σας συγχωρούμε για την ε, ανάληψη της Προεδρίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κίρκοπ. Ευχαριστώ κύριε Κίρκοπ. Ο κύριος Μπίσκι έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ένας γείτονας, ένας ένας γείτονάς μας, ένας Πολωνός, είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ ως ε, Ανατολικό Γερμανός ε, προέρχομαι από τη Σλούβιτσε, από την ε, Φραγκφούρτη Αντερόδε που είναι κοντά στη Σλούβιτσε και είναι αυτό ένα κομμάτι της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ευκαιρία να έλθει κοντά η Δυτική με την Ανατολική Ευρώπη ενώ έχουν μείνει χωριστά αυτά τα δύο κομμάτια της Ευρώπης για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλω να τονίσω και την ιδιαίτερη συμβολή της πολωνικής κουλτούρας στην Ευρώπη, την ε, ικανότητά σας να προωθήσετε τη συνεργασία και την διατήρηση της, πολιτικής, της πολιτιστικής πολυμορφίας. Εγώ έχω την τιμή να έχω δύο από τους γιους μου οι οποίοι μιλούν πολωνικά και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς Πολωνούς οι οποίοι συνέβαλαν πάρα πολύ στην πολωνική κουλτούρα και νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους η Ευρώπη να μην ξεχάσει τη μεγάλη συμβολή της Ανατολικής Ευρώπης μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο και θα έχετε την πλήρη μας υποστήριξη κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο πρόεδρος της ε, ε, Ευρω... Ο κύριος έχει το λόγο. Κύριε πρόεδρε, νομίζω σήμερα είναι ένα είδος ενθρονισμού. <clears throat> Είναι κρίμα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν πραγματικό κοινοβούλιο δεν επιλέγει επί τη βάση της ικανότητας τους προέδρους του και απλώς ακολουθεί τις αποφάσεις των πολιτικών ομάδων. Εμείς είχαμε στρατιώτες του Ευρωπαϊκού Στρατιωτικού Σώματος κυκλοφορώντας με την Ευρωπαϊκή Σημαία. Είχαμε ορχήστρα, χοροδίες κτλ. Ξεκινήσαμε σήμερα με τον Ευρωπαϊκό Ύμνο. Αλλά αυτός ο ύμνος δεν έπρεπε να υπάρχει από τη στιγμή που οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί είπαν όχι, και πολύ σωστά, στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή προωθείται όλα τα, τα σύμβολα μιας οντότητος, μιας κρατικής οντότητος και συγχρόνως προσπαθείτε να προσετεριστείτε τους Ιρλανδούς με εγγύησεις οι οποίες δεν αξίζουν τη μελάνη και το χαρτί πάνω στο οποίο έχουν γραφτεί. Εμεί, η ομάδα τη Ελευθερία και τη Δημοκρατία, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να υποστηρίξουμε το όχι στο Ιρλανδικό δημοψήφισμα, γιατί το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία εξακολουθεί να στηρίζεται στου ώμου των Ιρλανδών. Αγωνιστήκατε κατά τη Σοβιετική Ένωση, αγωνιστήκατε για τη δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε, αγωνιστήκατε για την εθνική ικανότητα αυτοδιάθεση. Αλλά εξακολουθείτε να αγνοείτε τη δημοκρατική φωνή χωρών όπω η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία, τότε αυτό θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένα είδο ένωση κατά τη οποία έχετε αγωνιστεί στο παρελθόν. Ακούστε πια τη φωνή των λαών. Ε, Ευχαριστούμε τον κύριο Φαράζ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις. Περί αυτού πρόκειται. Λίγοι λοιπόν ο γύρος των ομιλιών Βλέπω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, θα ήθελε και εκείνος το λόγο. Κύριε Μπαρόζο, έχετε το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, Ζέρσι Μπούζεκ, θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ προσωπικά και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκλογή σας στο ύπατο αξίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πολιτική σας πορεία υπέρ της ε, ελευθερίας δημοκρατίας και το γενικότερο σας θάρρος προώθησε τη θέση της χώρας σας, της Πολωνίας. Γίνατε πρωθυπουργός, ήσασταν πρωθυπουργός πριν ε, αναλάβετε το ρόλο του Ευρωβουλευτή. Προσπαθήσατε να προσεγγίσετε τις θέσεις της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης τις αξίες σας, τις οποίες υπερασπιζόσαστε. Και τώρα αναλαμβάνετε τα νέα σας καθήκοντα ως ε, πρόεδρος του Κοινοβουλίου. 20 χρόνια μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου, βλέπουμε ότι ζούμε μια επανενωμένη Ευρώπη. Εκτιμούμε την προσωπικότητά σας, το πολιτικό σας όραμα και τις μάχες που δώσατε. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να διαδραματίσετε έναν ενεργό ρόλο ως πρόεδρος υπέρ της Ευρώπης και των πολιτών. Η πείρα σας και οι αξίες αυτές θα οδηγήσουν σε μία ομαλή ε, ε, μετάβαση μεταξύ του Hans Gert Petering και ημών και τον οποίο θα ήθελα να συγχαρώ διότι κατάφερε να ανταποκριθεί στο καθήκοντα, στα καθήκοντά του αμερόληπτα. Και ενώπιον μιας δύσκολης πολιτικής στιγμής θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι για να προωθήσουμε την Ευρώπη. Οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου θα ενισχυθούν με τη συνθήκη της Λισαβόνας και πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου καθώς και η Επιτροπή θέλουν να εγκριθεί. Πρόκειται για μια συνθήκη που έχει εγκριθεί από 26 εθνικά κοινοβούλια και γι' αυτό θα πρέπει να την σέβονται όλοι οι ευρωβουλευτές. Τα θεσμικά μας όργανα θα ενισχυθούν και αυτό ισχύει και για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Γνωρίζουμε ότι μόνο με τη συνεργασία των δύο θεσμικών οργάνων θα προωθήσουμε την ε, ευρωπαϊκή υπόθεση. Γι' αυτό, Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, σας εύχομαι σε εσά καθώς και στο νέο κοινοβούλιο ε, πολύ καλή εργασία έτσι ώστε να προωθήσουμε τις ελευθερίες και την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκόλνης που εκπροσωπεί τους μη εγγεγραμμένου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι βέβαια ένας από τους μη εγγεγραμμένους. Θέλω εξ ονόματος τους να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου Βέβαια δεν σας συγχαίρω για τον τρόπο με τον οποίο εξελέγεστε, διότι, εξελέγετε, διότι αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με ένα τεχνητό τρόπο συνενώνονται για τις εκλογές του Πρόεδρου και μετά συνδιαχειρίζονται το Κοινοβούλιο για πέντε χρόνια. Ελπίζω λοιπόν κύριε Πρόεδρε να ξεπεράσετε αυτή τη νίκη, να μην είσαστε ο σκλάβος των δύο αυτών μεγάλων πολιτικών ομάδων, να μπορέσετε να υποστηρίξετε και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των μειοψηφιών και ιδίως των αντιφρονούντων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτών οι οποίοι ανησυχούν για τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στον οικονομικό κλάδο για το κίνδυνο να χάσουμε την ταυτότητά μας, για την ανάμιξη των προσώπων, των κεφαλαίων, των εμπορευμάτων δεν νομίζουμε ότι από αυτά θα προέλθει οτιδήποτε το καλό και που είναι εναντίον της ατέρμονης αύξησης των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί των εθνικών εξουσιών. Είμαστε οι αντιφρονούντες που υπήρξετε και εσείς ο ίδιος αντιφρονών στο παρελθόν. Ελπίζω θα προστατεύσετε τα δικαιώματά μας και ιδίως, ιδίως ότι θα σεβαστείτε τον κανονισμό αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος δεν πρέπει να το τοποποιείτε συνέχεια όταν αντιλαμβάνονται ορισμένοι ότι μπορούν να ευνοηθούν αυτοί που δεν θέλουν την πραγματικά ελεύθερη έκφραση των ευρωπαϊκών λαών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όσα είχατε να πείτε. Εξ τον των μη γεγραμμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα τώρα να σας ανακοινώσω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτό το τμήμα της συνεδρίασης και εξαντλούμε και το σημείο της διάταξης εκλογή του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα περάσουμε τώρα στην εκλογή των αντιπρόεδρων. Όσον αφορά την εκλογή των αντιπρόεδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνω να ορίσουμε μία προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιωτήτων για τις μία το μεσημέρι. Μία το μεσημέρι είναι η προθεσμία. Ελπι... περακαλώ